Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας με μεγάλη χαρά. Καλωσορίζουμε το φίλο μας, τολμώ να πω φίλο μας, γιατί είναι η τρίτη φορά που παρίσταται στις εργασίες μας, τον Υπουργό Αντώνιο Μιλοσοευσκή, Υπουργό Εξωτερικών και θα το πω πρώτη φορά και τελευταία με το πλήρες όνομα, πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και μετά θα λέω Μακεδονία, με την ελπίδα ότι θα λυθεί και το πρόβλημα του ονόματος, λέγει ο Πρόεδρος. Γνωρίζετε κύριε Υπουργέ το ενδιαφέρον που το Κοινοβούλιο αλλά και η Επιτροπή μας για τις εξωτερικές υποθέσεις ε, παρακολουθεί, το ενδιαφέρον με το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις ε, στη χώρα σας που οδηγούν προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έγιναν προεδρικές εκλογές το Μάρτιο, διοικητικές τον Απρίλιο και ο τρόπος με τον οποίο εκτιλήχθησαν οι εκλογές ήταν κοινή ομολογία επιτυχής και δημοκρατικός. Έγιναν, σημειώθηκαν σημαντικές πρόοδοι. Κάτι το οποίο αποτελεί και ουσιώδες κριτήριο, ουσιώδη παράγοντα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρόοδοι αυτές μεταφράστηκαν και στην αναφορά της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ζητεί και συστήνει έναρξη των διαπραγματεύσεων. Για αυτούς τους λόγους και η Επιτροπή μας προσφάτως εξέφρασε την πριν της υποστήριξη στην κατάργηση των θεωρήσεων για τους Μακεδόνες υπηκόους. Το υποσχέθηκε ο πρόεδρος όταν λέει Μακεδονία τη χώρα και Μακεδόνες τους κατοίκους. Και ας ελπίσουμε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει από πρώτης πρώτου του επομένου έτους. Τώρα, Υπάρχει και το πρόβλημα, το βάζω εντό εισαγωγικών γιατί δεν είναι και τόσο σοβαρό πιστεύω, του ονόματος που θα μπορούσε ενδεχομένω να αποτελέσει εμπόδιο στην εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Είναι όμως σημαντικό να εξευρεθεί συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση επί του θέματος της ονομασίας για να τεθεί ένα οριστικό τέλος στην αντιπαραγωγική αυτή αντιπαράθεση. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες προκλήσεις που αναμένουν την Μακεδονία πριν επιτυχεί το στόχο της ε, ένταξης κατά πολέμηση της διαφθοράς, μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, ενίσχυση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας της, μεταρρύθμιση στην εθνική διοίκηση, σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, πολλά και διάφορα πρέπει να γίνουν. Βλέπουμε όμως μια ειλικρινή διάθεση και αποφασιστικότητα εκ μέρου των μακεδονικών αρχών να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά. Δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στον Υπουργό και μετά στους συναδέρφους για να ακολουθήσει ένας ελπίζω και είμαι σίγουρος ενδιαφέρον διάλογος. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την άδειά σας στον οίκο αυτών όλων των ευρωπαϊκών εθνών μεγάλων και μικρών θα σας παρουσιάσω την ομιλία μου στην μητρική μου γλώσσα τα μακεδονικά έτσι ώστε να συνεισφέρω και εγώ στον εμπλουτισμό του ευρωπαϊκού πολυπολιτιστικού φάσματος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και την πρόσκλησή σας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι για μένα είναι τιμή αυτή η ομιλία ενώπιον της Επιτροπής σας για πρώτη φορά μετά από τις ε, τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές ε, τον Ιούνιο. Πάντα με χαρά συναντούσα τα μέλη της Επιτροπής σας, γιατί τέτοιες συναντήσεις μας δίνουν την ευκαιρία να σκεφτούμε επικοδομητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Είμαι πεπισμένος ότι θα υποφελθούμε από αυτή την ευκαιρία για να δούμε τι πρόοδος έχει γίνει στη Μακεδονία και ποιες είναι οι δυνατότητες για περαιτέρω πρόοδο στον δρόμο προς την Ένωση. Οι προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες και θα τις συμπεριλάβουμε στον οδικό χάρτη που θέλουμε να καταρτήσουμε στο δρόμο της Μακεδονίας για την ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Με την ίδια ευκαιρία σας συγχαίρω για την κατάληξη της διαδικασίας επικύρωσης της Λισαβόνας που είναι τόσο ουσιώδης για να συνεχιστεί η διαδικασία της διεύρυνσης. Σήμερα η Δημοκρατία της Μακεδονίας αντιμετωπίζει μια αποφασιστική καμπή. Η δυνατότητα αρχής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων είναι μπροστά μας η δυνατότητα να επεκταθεί δηλαδή η ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και ασφαλείας στην Ευρώπη 20 χρόνια μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου είναι και αυτή κάτι το εφικτό. Η δυνατότητα η μικρή και φιλιρινική χώρα της Μακεδονίας να εισέλθει στην ευρωπαϊκή οικογένεια εθνών είναι τώρα πια πραγματικότητα. Η ευθύνη είναι κατά πρώτον λόγο δική μας, δηλαδή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και όλων των πολιτικών παραγόντων στη χώρα. Αλλά είναι και, και κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και δική σας και δική μας. Για να διασφαλίσουμε την ευημερία των τωρινών και μελλοντικών γενεών των πολιτών της Μακεδονίας με την εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων, η κυβέρνηση δίνει την ύψιστη προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας μας. Εφόσον αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος όλων των κυβερνήσεων από την ανεξαρτησία το 1991 μέχρι σήμερα. Και το στόχο αυτό συμμερίζονται όλοι οι πολίτες και εθνοτικές κοινότητες καθώς και πολιτικά κόμματα δημοσκόπηση έδειχνε ότι 90% των πολιτών της Μακεδονίας υποστηρίζουν την ολοκλήρωση, τη συμπερίληψη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλων των χωρών του Συμφώνου Σταθερότητας γιατί αυτό είναι και τμήμα της, ε, του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Όπως ξέρετε πριν από μερικές εβδομάδες η Κομισιόν έκανε μια αξιολόγηση των προόδων της Μακεδονίας προς την ένταξη και ο βαθμός εκπλήρωσης των κριτηρίων ένταξης που καθόρισε η Ένωση ήταν τόσο ικανοποιητικός ώστε μπορούν ίσως να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την υποστήριξη βέβαια του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν καθώς και όλων των χωρών μελών. Επίσης πρέπει να τονίσω ότι η συνένεση μεταξύ των κομμάτων ως προς το στόχο αυτό είναι επίσης ουσιώδης. Η υποστήριξή σας ήταν πολύ ευπρόσδεκτη και ελπίζω να συνεχιστεί και στο μέλλον. Επίσης με χαρά διαπιστώνω ότι ο εισηγητής κύριος Ζόραν Τάλερ σημείωσε τα επιτεύγματα αυτά στην έκθεση που εξετάσατε την περασμένη εβδομάδα και με αυτή την ευκαιρία θέλω να εκφράσω όλη μου την εκτίμηση για την υποστήριξη αυτή και την μελλοντική υποστήριξη που αναμένουμε για το επόμενο ψήφισμα, την αρχή δηλαδή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αλλά και της πλήρωσης ορισμένων χασμάτων και ελλείψεων. Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ γιατί πρέπει να αναλάβουμε και να εφαρμόσουμε πολλές μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχει ήδη αναλύσει και προβλέψει η κυβέρνηση και πάνω σε αυτές θα βασιστούν όλα μας τα μελλοντικά προγράμματα. Έχουν ήδη μεταφραστεί σε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις συστάσεις της Ένωσης. Θα είναι επίσης η βάση για την τακτική ετήσια αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει μεταρρυθμίσεις και ελπίζουμε να καταλήξει σε αυτά αποτελέσματα για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και κριτηρίων επιμείνουμε στη μεταρρύθμιση της κρατικής διοίκησης του δικαστικού συστήματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας, της εφαρμογής της Συμφωνίας Πλαισίου της Αχρίδας, της επίτευξης των, εφαρμογής μάλλον των υποχρεώσεών μας με βάση στα πλαίσια της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Ένταξης και επίσης την κοινωνική πολιτική, τον ενεργειακό τομέα κλπ. Η κυβέρνηση επίσης έχει υποσχεθεί να επιτύχει πρόοδο στις σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει αυτή η διαμάχη με την Ελλάδα για το όνομα και συνεχίζουμε με αυξημένη δυναμική να προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για μια αμοιβαία αποδεκτή συνθήκη που να μην βλάπτει το γόητρο του μακεδονικού λαού. Θέλουμε και θα έχουμε άμεσες επαφές με τους Έλληνες συναδέλφους μας με ανοιχτό πνεύμα σύμφωνα με το πρότυπο των συνεννοήσεων Κροατίας και Σλοβενίας. Και νομίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να λύσουμε το μόνο διμερές ανοιχτό πρόβλημα που έχουμε. Η Μακεδονία πιστεύει ότι πρέπει να έχει φιλικές σχέσεις με όλες τις γειτονικές της χώρες. Και αυτό φαίνεται και από τη διευθέτηση των συνοριακών θεμάτων με το Κωσυφοπαίδιο, πράγμα που συνεισφέρει στην αύξηση της περιφερειακής ασφάλειας σε όλες τις περιφερειακές μας πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την απελευθέρωση του στο θέμα των θεωρήσεων. Νομίζουμε ότι η Μακεδονία θα δείξει το ίδιο ανοιχτό πνεύμα με την ίδια την Ένωση με βάση τις αρχές της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας και ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών. Πιστεύουμε ότι μετά της, ε, την καινούργια κυβέρνηση στην Ελλάδα μετά τις τελευταίες εκλογές μπορεί να βελτιωθεί το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών και το πρόβλημα της ονομασίας. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε σημαντική πρόοδο γιατί η Μακεδονία αναμένει αποτελέσματα και οι προσπάθειες που έχουν γίνει για την βελτίωση των σχέσεων δεν περιορίζεται στην Ελλάδα και το όνομα αλλά σε όλες τις γειτονικέ χώρες και νομίζουμε ότι αυτό θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο τέλος του έτους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί τελικά να πετύχει πολιτική συμφωνία και να ζητήσει επίσημα την αρχή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Πράγμα που θα ήταν σημαντικό και για την ε, διαδικασία σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβεβαιώσει την αξιοπιστία της ε, διαδικασίας διεύρυνσης που έχει δεχτεί. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από το ρυθμό και την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων και θα οδηγήσει με τη σειρά του σε άλλες οικονομικού τύπου μεταρρυθμίσεις και στις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση της σταθεροποίησης στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οποιαδήποτε δε καθυστέρηση θα έχει αποθαρρυντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές που θα ήθελαν η Μακεδονία να είναι ένα σύγχρονο κράτος μέσα στην Ευρώπη με έκφραση όλων όλου του δυναμικού της και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία θα ενδυνάμωναν και τις ε, σχέσεις μεταξύ μειονοτήτων στη Μακεδονία, γιατί είναι πολυεθνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα να σας πω μερικά και για το θέμα των θεωρήσεων, που είναι από τους σημαντικότερους στόχους της κυβέρνησής μας για φέτος. Ο καθορισ... Ε, η απελευθέρωση των θεωρήσεων για ταξίδια στην Ένωση είναι σημαντικό θέμα και για τους πολίτες της Μακεδονίας και για τους πολίτες άλλων χωρών της περιοχής μας. Η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες να πληρώσει όλα τα κριτήρια που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αδικασία κοντεύει να λήξει και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της, την υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης της Κομισιόν για την κατάργηση των θεωρήσεων. Πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει μεγαλύτερη συνεργασία πιο ευκολότερη μεταξύ Μακεδονίας και Ευρωπαίων πολιτών και θα δώσει την ευκαιρία στους νέους να μάθουν πολλά πράγματα επισκεπτόμενοι τις ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τη σημαντική λοιπόν σημασία που έχει η κατάργηση των θεωρήσεων, δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν υποκατάστατο για τις ίδιες τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Είναι ένα απλό εργαλείο για την ένταξη, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός. Η κατάργηση των θεωρήσεων ήταν κάτι πολύ θετικό για τη Μακεδονία γιατί έδειξε ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα πολύπλοκα τεχνικά κριτήρια που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προϊονίζει θετικά τις, διαπραγματε... τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Έχουμε δυνατότητες και θα τις χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται από την αρχή των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το θέμα του προενταξιακού εργαλείου που είναι και για, για μας επίσης σημαντικό. Η πλήρη χρησιμοποίηση των κονδυλίων που μας χορήγησε η Ένωση είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για την κυβέρνησή μας. Ένας από τους στόχους στο πλαίσιο αυτό είναι η αποκεντρωμένη χρησιμοποίηση των κονδυλίων αυτών μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και στην θεσμική προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή του εργαλείου αυτού, του προενταξιακού εργαλείου. Έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες απορρόφησης και αυτό φαίνεται από την από τον τρίτο του πυλώνα την περιφερειακή ανάπτυξη και τον τέταρτο τη χρησιμοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Σύντομα θα σας πω μερικά για τη γενικότερη οικονομική κατάσταση. Η γενική οικονομική κρίση σημειώθηκε και στη Μακεδονία. Ακυρώθηκαν παραγγελίες στον μεταλλουργικό και υφαντουργικό τομέα. Αλλά η Μακεδονία αποτελεί τελικά θετικό παράδειγμα όχι μόνο για την περιοχή της αλλά και γενικότερα. Η πτώση του ΑΕΠ στη Μακεδονία ήταν μόνο 1,2% ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε κατά 0,4% τους πρώτους 9 μήνες του 2009. Η κυβέρνηση κατάφερε μάλιστα να διατηρήσει το έλλειμμα μέσα στα πλαίσια του 2,8% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα και η ανεργία δεν ήταν τραγικών διαστάσεων. Οι βασική λόγοι για αυτή τη μικρή μείωση του ΑΕΠ είναι η ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση, τα χαμηλά επιτόκια, η ψηλή οτσεκούβαμε μαλ Αποταμίευση και η αύξηση του ΑΕΠ το τέταρτο, κατά το τέταρτο τμήμα του 2009 προβλέπεται να είναι χαμηλή μένα αλλά μόνο κατά 0,6% χαμηλότερη. Χάρη σε ορισμένα μέτρα της κυβέρνησης όπως το, τη φορολογική δέσμη που αφορούσε τους φόρους που οφείλονταν από εταιρείε και μια δέσμη 70 μέτρων κατά της κρίσης μεταξύ των οποίων υποστήριξη δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για επιχειρήσεις και διευκολύνσεις για, τη διαχείριση μιας, για την ίδρυση επιχειρήσεων στη χώρα. Κυρίες και κύριοι βουλευτέ, έχω έρθει σήμερα, ήρθα σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα της ε, ε, μακεδονικής ένταξης. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε καλά πόσο εκτιμούμε το διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήρθα όμως επίσης να ζητήσω την υποστήριξή σας για την επόμενη φάση του δρόμου προς την Ένωση, δηλαδή το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Οι Μακεδόνες θεωρούσαν πάντοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ένα φάρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ελπίδας και σήμερα προσβλέπουν σε ισχυρή υποστήριξή σας για την αρχή των διαπραγματεύσεων. Έχουν σημειωθεί κοινέ επενδύσεις σε σημαντικά πολιτικά και οικονομικά κεφάλαια, γι' αυτό και τώρα πρέπει από κοινού να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η προσδοκία των πολιτών της χώρας μου είναι να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις του χρόνου. Το 2010 θεωρείται ως έτος νέας αρχής, στην οποία θα γιορτάσουμε την εκατοστή επέτειο από τη γέννηση της μητέρας Τερέζας. Και επιτρέψτε μου τώρα να καταλήξω με μία σκέψη της ανθρωπίστριας αυτής. Που είπε, θεωρούμε ότι το, αυτά που κάνουμε είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά ο ωκεανός θα ήταν λιγότερος αν έλειπε η σταγόνα αυτή. Λιγότερο σημαντικός. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας και το 2010 εύχομαι να αρχίζουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Το έχω ξαναπεί. E Πριν ξεκινήσουμε αυτή καθ' αυτή ε, συζήτησή μας, θα δώσω το λόγο για τέσσερα λεπτά στον συνάδελφο Τάλερ, που είναι εισηγητής για το θέμα της ένταξης της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέσσερα λεπτά, κύριε Τάλερ. Ευχαριστώ κύριε Αλμπερτίνη. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για την ε, επικοδομητική ε, ομιλία σας και ε, για τη διαλλακτική σας θέση. Νομίζω ότι είναι καλό για την ε, ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει εδώ στην ε, Επιτροπή. Η συνάντηση την οποία είχαμε με έχει, μου έχει επιβεβαιώσει την εντύπωση ότι συμπεριφέρεστε πολύ καλά σαν Υπουργός Εξωτερικών, σαν πολιτικός και ε, συμβάλλεται ε, η ΦΥΡΟΜ να μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το, το έτος αυτό ήταν πολύ καλό για τη χώρα σας στις 19 Δεκεμβρίου θα απελευθερωθούν οι θεωρήσεις και ε, έχουμε την έκθεση με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιλύσατε και τη σχέση σας με το κοσυφοπέδιο, άρα έχετε πολύ καλά επιτεύγματα. Οπότε αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μπορέσουμε να έχουμε μία πραγματική πρόοδο ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ΦΥΡΟΜ ε, προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλα αυτά τα χαιρετίζω και πιστεύω ότι θα πρέπει να βρείτε και μία λύση με τη γειτονική σας χώρα την Ελλάδα ότι θα πρέπει να λύσετε και τη διμερή διαφωνία σας ως προς την ονομασία θα δείτε ότι οι συνάδελφοι θα κάνουν ερωτήσεις και αυτό το θέμα θα απασχολήσει πολλές ερωτήσεις διότι αναρωτιέται κανείς γιατί έχετε τόσο λίγες σχέσεις με την γείτονα χώρα. Αλλά εδώ ε, είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, είμαστε πλειοψηφικά υπέρ της ε, προσχώρησης της ΦΥΡΟΜ και συζητάμε και με τους Έλληνες συναδέλφου μας. Πιστεύουμε ότι έχει ανοίξει ένα παράθυρο, μια ευκαιρία και θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται. Θα ήθελα εδώ να σας πω ότι ε, αντιλαμβάνομαι ότι είχατε μία ιστορική συνάντηση με τον κύριο Παπανδρέου τέλη Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, πράγμα το οποίο μπορεί να είναι η απαρχή αμοιβαίου σεβασμού και θα πρέπει τώρα να προσπαθήσουμε να βρούμε ε, ε, μία συμβιβαστική λύση. Ως εισηγητής έχω ένα όνειρο. Ε, ε, και οι άλλοι, ε, και άλλες γειτονικές χώρες η Ελλάδα και η Βουλγαρία να στηρίξουν την προσχώρηση της ΦΥΡΟΜ διότι είναι πολύ βασικό για μας να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα όνειρά μας το όνειρο το οποίο έχει και ο κύριος Παπανδρέου δηλαδή η ΦΥΡΟΜ να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ τον κύριο κύριο Τάλ. Πριν αρχίσει η συζήτηση, θα μιλήσει ο κύριος Αλαφράγκα από το πιο πολυπληθές κόμμα το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Υπουργού και να τον ευχαριστήσω για την απόλυτη και πάγια διάθεσή του ε, να έχει διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, ο διάλογος για την επίλυση των εκκρεμών προβλήματων. Και μπορώ να σας πω κύριε Υπουργέ ότι και εμείς διαβάσαμε μεγάλη προσοχή την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πρόοδους που έχει επιτελέσει η χώρα σας και στο όνομα της πολιτικής μου ομάδος μπορώ να σας πω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτές τις πρόοδους. Ιδιαίτερα, σε τη συνένεση των διαφόρων πολιτικών δυνάμεων, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για το νομοσχέδιο χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, για τη λειτουργία του, Ευρωπαϊκού ε, του Εθνικού Κοινοβουλίου, για την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Οι πρόοδοι είναι λοιπόν πολύ σημαντικές και αξιοσημείωτες και γι' αυτό θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη διάθεση της κυβερνήσεώς σας να συμμετάσχει και στις αστικές πολιτικές αλλά και στρατιωτικές επιχειρήσεις που η ε, Ευρώπη έχει ανά τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το βασικό σημείο το οποίο τόλισε και ο εισηγητής και μάλιστα αποφασιστήκα είναι η επίλυση του τελευταίου ε, εκκρεμούς προβλήματος. Θα ήταν ιδιαίτερα λοιπόν παρά και μετά την επίλυση όλων των λοιπόν ουσιαστικά προβλημάτων και την πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα ε, που της δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις να προσκρούσει πάλι στο τείχος, στο εμπόδιο ενός θέματος που δεν αφορά την ουσία ουσιαστικά επιτρέψατε μου να πω που δεν είναι ουσιαστικό Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι αναμένουμε και εμείς ελπίζουμε σε μία να τον ταχύτερη λύση για να μπορέσουμε και επισήμως να γιορτάσουμε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει όμως να ανασκουμποθούμε όλοι για να εξεύρουμε λύση στο τελευταίο, επαναλαμβάνω, εμπόδιο που υπελείπεται και που ορθώνεται στο δρόμο της ε, φύρων προς την ε, ένταξη. Το ερώτημά μου, υπό το φως των νέων δυνατοτήτων ε, που ανοίγει η ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προοπτικές για την υπερπίδηση αυτού του τελευταίου εκκρεμούς προβλήματος. Έχοντας κατά νου ότι δεν είναι το ουσιαστικό ναι. πρόβλημα. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα ουσίας. Ευχαριστώ κύριε Σαλαφράγκα. Κάτσιν, δύο λεπτά παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο. Ευχαριστώ. Spoštovani gospod minister, iskrene čestitke za... Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για την επιτυχία στην οδό προς την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τη χώρα σας και τη Βοσνία Ερζεγονιβίνη. Η Φύρομ μπόρεσε όντως να εκπληρώσει το στόχο αυτό, τα κατάφερε πιο γρήγορα από ό,τι παραδείγματο χάρη το Μαυροβούνιο και μπόρεσε να αποτελέσει μια κινητήριο δύναμη για να προωθηθεί το θέμα της κατάργησης των θεωρήσεων. Σας ε, συγχαίρω και ελπίζω ότι η χώρα σας θα βοηθήσει την Αλβανία και το Κωσυφοπέδιο ε, διότι το Κωσυφοπέδιο δεν έχει καν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και η Αλβανία είναι γειτονά σας. Ε, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τις θεωρήσεις ήδη στις 19 Δεκεμβρίου πριν την χρονιά. Αυτή είναι η πρόταση της χώρας μας και της Υπουργού μας Εξωτερικών της χώρας από την οποία προέρχομαι. Ε, βεβαίως ε, το δικό σας ε, κράτος περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις οπότε εγώ θα απέφευγα να καθορίσουμε ημερομηνίες αλλά έχετε κάνει μεγάλες προόδου, ιδίως διότι το κοσυφοπέδιο δεν πάει καλά η, Βοσνη, η βοσνιακή κοινότητα θεωρείται ότι απειλεί, θεωρεί ότι απειλείται ε, έχουμε υπερψηφίσει το ψήφισμα της Ρεμπενίτσα, κάτι το οποίο θεωρούμε ότι έπρεπε να γίνει. Το έκανε η, το Ζάγκρεπ, το έκανε η Προκορνίτσα και καλό θα ήταν να το πράξετε κι εσείς, ε, διότι δεν θέλουμε απλούστατα να ξεκινήσει η χώρα σας, αλλά να μπορέσει να αποτελέσει κινητήριο δύναμη κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαπραγματεύσεις και με το κοσυφοπέδιο. Ευχαριστώ κύριε Κάτσινγκ. Ο κύριος Στάνοκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Καταρχήν, εν ονόματι της ομάδας μου των Άγγλων Συντηρητικών θα ήθελα να σας συγχαρώ διότι προχωράτε στην επόμενη φάση σαν υποψήφοι για να διαπραγματευτείτε την προσχώρησή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Όσον αφορά την καταπολέμηση της εγκληματικότητος και της διαφθοράς έχετε κάνει προόδους, το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις και ελπίζω ότι τώρα η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να σας δώσει το πράσινο φως για τις πρώτες συζητήσεις. Πάντως συνεχίζει το θέμα της ονομασίας με τον όρο φύρομ και η ελληνική κυβέρνηση ε, διαφωνεί παρόλο που η νέα κυβέρνηση είναι πιο ευέλικτη. Ε, στη χώρα μου ε, αντιλαμβάνομαι ότι η Μασεντόνια έχει βλέψεις προς τη Μακεδονία. Για μένα πρόκειται για ένα μύθο ε, εχθρικές ε, προθέσεις εκ της χώρας σας προς την γείτονά σας. Μπορείτε να επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να ε, αρνηθείτε κατηγορηματικά και να πείτε ότι δεν έχετε καμία βλέψη προς τη γείτονα χώρα σας και να γνωρίζετε τα σύνορά σας ως τελεσίδικα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κούκαντ για δύο λεπτά. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ε, χαιρετήσω τον Υπουργό, να τον ευχαριστήσω για τα σχόλιά του. Είναι όντως μεγάλη χαρά διότι από τη χώρα σας ε, έχουμε τόσο θετικά νέα τα, τους τελευταίους μήνες. Θα συζητήσαμε τελευταίως, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Πρόκειται για την ικανοποίηση όλων των κριτηρίων, για την κατάργηση του συστήματος θεωρήσεων ε, και ε, για την εκπλήρωση των στόχων της Κοπενχάγης όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια που θα επιτρέψουν το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Είναι όντως θετικά νέα που πρέπει να ενθαρρύνουν την κυβέρνησή σας να εντείνει τις προσχάθειές της σε αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν ε, καθορίζεται την, ε, ε, ότι θα καθοριστεί όπου να είναι η ημερομηνία διότι σε λίγες μέρες θα ολοκληρώσουμε τέσσερα χρόνια που είναι η χώρα σας υποψήφια και το Δεκέμβριο το Συμβούλιο θα επιτρέψει να ξεκινήσουν στο δυνατόν πιο γρήγορα οι διαπραγματεύσεις. Για τις επιτυχίες ε, μίλησαν οι συνάδελφοι ήδη. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυβέρνηση στην, ε, ε, στη Φύρομ είναι τέτοια ώστε η κυβέρνηση Γκρουεύσκη είναι καλά εγκατεστημένη εκλεγμένη στη χώρα και μπορεί να χρησιμοποιήσει την ε, θέση της για να ηγηθεί. Δηλαδή η κυβέρνηση θα έπρεπε να αναλάβει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον. Πράγμα το οποίο θα επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να επιλύσει όλα τα ουσιαστικά προβλήματα. Καλό θα ήταν αν μπορέσετε να συνεχίσετε τέτοιες πρωτοβουλίες και να τις εφαρμόσετε και στο θέμα του ονόματος. Ευχαριστώ τον κύριο Κούκαν. Το λόγο έχει η κυρία Κοπά για δύο λεπτά. Θέλω να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών και πάντα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ανταλλαγή απόψεων όσες φορές έχει έρθει. Ε, θέλουμε και εμείς να χαιρετήσουμε την πρόοδο της χώρας που είναι σημαντική για όλα συνολικά τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπάρχουν όμως ακόμα ανοιχτά ζητήματα. Και όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα σε αυτή την Επιτροπή και όπως έχει αποδείξει η εμπειρία της Κροατίας σε σχέση με τη Σλοβενία, ο δρόμος της Ευρωπαϊκής, για την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από τη διευθέτηση των προβλημάτων που αφορούν την καλή γειτονία. Και αυτό καλείται σήμερα η χώρα να ε, λύσει. Από πλευρά τη Ελλάδα, μετά τις εκλογές, είναι καθαρή επιθυμία της νέας κυβέρνησης να προχωρήσουμε με γρήγορο ρυθμό στο διάλογο για το μόνο θέμα που μας χωρίζει, δηλαδή για μια κοινά αποδεκτή ε, ονομασία. Και η συνάντηση πράγματι Παπαντρέου Γκρούευσκη ήταν ένα πολύ καλό σήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Η ελληνική θέση είναι σαφής, σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό που διαφοροποιεί τη χώρα από την γεωγραφική Μακεδονία, έργα όμνης. Για μας το πλαίσιο παραμένει το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, από την άλλη, ο πολλαπλασιασμός των επαφών είναι πάντα θετική, θετικός και γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις για συζήτηση ώστε να πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Το κρίσιμο όμω θέμα το οποίο κύριε Υπουργέ θέλω να θέσω είναι το ζήτημα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών στην περιοχή μας και όχι μόνο μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας σας αλλά και σε σχέ... ανάμεσα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τη Βουλγαρία. Και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης είναι η βάση για να λυθούν όλα τα άλλα θέματα στην περιοχή. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι έχει σκοπό η κυβέρνησή σας με τη σημερινή συγκυρία, με τη δεδομένη τοποθέτηση της Επιτροπής, με τη νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες όχι μόνο σχετικά με το όνομα, αλλά και με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης συνολικά για την περιοχή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για δύο λεπτά η Μπρίζετσικ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας συγχαρώ για τις επιτυχίες που σημειώθηκαν και που αναφέρονται στην έκθεση της Κομισιόν. Δέχεστε ότι υπάρχουν ακόμη ελλείψεις μεταξύ των οποίων το ότι μεταξύ των επιτυχιών μάλλον η επίλυση των, διαμεθοριακών, των μεθοριακών προβλημάτων με το κοσυφοπέδιο. Πράγματι αυτά είναι δύσκολα προβλήματα σε χώρες όπως των Βαλκανίων. Ερωτώ λοιπόν, Έχετε κανένα άλλο θετικό πρόγραμμα ή σχέδιο ή πρωτοβουλία για βελτίωση των σχέσεών σας με το κοσυφοπέδιο, περαιτέρω βελτίωση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων και να ξαναπάρει το λόγο ο Υπουργός για απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όπως πρέπει. Ευχαριστώ και τον κύριο Τάλερ για όσα είπε. Από τη θέση του ως ηγητού όπως γνωρίζετε. Θα απαντήσω τώρα. Πρώτα του κυρίου Σαλαφράνκα, του σεβαστού μου κυρίου Σαλαφράνκα. Οι διαπραγματεύσεις με τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για επαφές, ανταλλαγές απόψεων και για την κατάστρωση κοινών σχεδίων για όλα τα θέματα που μπορεί να είναι κοινού ενδιαφέροντος, όχι μόνο για την ονομασία. Κυρία Κόπα, για ανάλογη ερώτηση. Αν έχουμε σχέδια δηλαδή για σχέδια οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή τίποτε άλλο που να μας φέρει πιο κοντά και να βοηθήσει αυτό έτσι τις σχέσεις καλής γειτονίας. Απαντώ θετικά και Νομίζω ότι πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα σε άμεσες επαφές. Έχουμε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση και το άνοιγμα νέων μεθοριακών σταθμών κοντά στις πρέσπες. Μάρκο Βανόγκα και Άγιος Γερμανός στα ελληνικά. Νομίζω ότι με τέτοια συγκεκριμένα θέματα, ε, τέτοιες συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα μπορούν όντως να μπορεί όντως να οικοδομηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Είναι μικρά βήματα αλλά σημαντικά για τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων. Και η δεύτερη πρωτοβουλία πριν από μερικές μέρες ο Υπουργός Οικονομικών της Μακεδονίας και εγώ ο ίδιος στείλαμε επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών και Πρωθυπουργό της Ελλάδος κύριο Παπανδρέου για να αρχίσουν, προτείνοντας να αρχίσουν συνεννοήσεις για να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση, διότι η ελληνική επιχειρησιακή κοινότητα είναι από τις μεγαλύτερες στη δημοκρατία της Μακεδονίας και εκείνοι είχαν ζητήσει οι δύο χώρες να υπογράψουν μια συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης ώστε να έχουν καλύτερες δυνατότητες ε, εμπορικών συναλλαγών στη Μακεδονία. Τώρα, οι ερωτήσει του κύριου Κάτσιν για τις θεωρήσεις. Θα ήθελα να σας πω ότι η Μακεδονία είναι διατεθειμένη να μοιραστεί την εμπειρία της και με την Αλβανία και με το Κωσυφοπαίδιο και τα επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα της κατάργησης των θεωρήσεων ή της απελευθέρωσης των θεωρήσεων γιατί οι Αλβανοί είναι μεν ε, πλειοψηφία στο Κωσυφοπέδιο και την Αλβανία, στη Μακεδονία όμως μειοψηφία, αλλά οι Μακεδονοαλβανοί θα είναι οι πρώτοι Αλβανοί των Βαλκανίων που θα έχουν το δικαίωμα να ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς θεώρηση. Αυτό είναι συμβολικό μέτρο για την πολυεθνική μας κοινωνία. Τώρα για το ψήφισμα για τη Ρεμπρένιτσα της Μακεδονικής Εθνοσυνέλευσης. Σας καλώ να, την, να το διαβάσετε και να προσέξετε ιδιαίτερα ότι η μακεδονική κυβέρνηση θα ήθελε να καταδικάσει μαζί με τον υπόλοιπο δημοκρατικό κόσμο τις σφαγές στην Σρεμπρένιτσα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το θυμούνται όλοι οι πολιτικοί της περιοχής μας για να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις στο μέλλον. Επίσης θα ήθελα να σχολιάσω το συγκεκριμένο ερώτημα του κυρίου Τάνοκ για τις ανησυχίες ορισμένων Ελλήνων για επεκτατικές μας τάσεις. Θα σας πω μερικά πράγματα. Πρώτον, η Μακεδονία είναι η μόνη χώρα στην περιοχή μας που στο σύνταγμά της έχει σαφώς δηλώσει ότι δεν έχει καμία εδαφική διεκδίκηση από καμία γειτονική της χώρα. Και αυτό το σέβονται όλοι οι πολιτικοί παράγοντες στη δημοκρατία της Μακεδονίας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σαφές και συγκεκριμένο όσον αφορά ακριβώς την εδαφική ακεραιότητα όλων των κυριάρχων κρατών της περιοχής. Η Μακεδονία, επαναλαμβάνω, είναι η μόνη χώρα από τη Σλοβενία μέχρι την Κύπρο που έχει καθορίσει τόσο σαφώς και τόσο ειρηνικά τα σύνορά της με όλους τους γειτονές της. Και αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι που δείχνει ότι δεν έχουμε καμία επεκτατική διάθεση προς κανέναν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι τα τελευταία 19 χρόνια από τότε που είμαστε ανεξάρτητοι δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ ούτε ένα θέμα παραβίασης ασφαλείας ή ατυχήματος σε σχέση με θέματα ασφαλείας με την Ελλάδα. Εκτός αυτού, Μακεδόνες και Έλληνες στρατιώτες συνεργάζονται στην ειρηνευτική αποστολή στο Αφγανιστάν, όπου η Μακεδονία έχει αποστείλει 3 περίπου τις 100 των στρατευμάτων της. Η προσωπική μου πεποίθηση και όλων των λογικών ανθρώπων νομίζω είναι ότι η ύπαρξη μίας ενιαίας και κυρίαρχης χώρας, κράτους όπως η Μακεδονία, δεν αποτελεί απειλή αλλά εγγύηση για τους Έλληνες γειτονές μας. Τέλος, να σας πω και ένα ανέκδοτο μεταξύ όλων αυτών των σοβαρών. Η Μακεδονία γενικά έχει 8 ελικόπτερα συνολικά και δύο είναι δωρεά της Ελλάδας και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Για να απαντήσω τώρα στο ερώτημα του κυρίου Κούκαν, ευχαριστώ πολύ. Και η απάντησή μου θα είναι θετική. Μάλιστα, σχεδιάζουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια χρηματοδότηση που διαθέτουμε για μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε πρόοδο και να επενδύσουμε όλες μας τις δυνατότητες για αποδοτικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στην οικονομία, σε στρατιωτική μεταρρύθμιση και σε καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Θέλουμε ως καινούργοι στην πολιτική την, δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κράτος. Τέλος, για να απαντήσω και στο ερώτημα της κυρίας Ιμπρεζάγκετς για το Κωσυφοπέδιο, η Μακεδονία αναγνώρισε την εξαρτησία του Κωσυφοπεδίου, καθορίσαμε τα σύνορά μας Πρόσφατα ήρθε και ο συνάδελφός μου από την Πρίστινα να μας επισκεφθεί επισήμως και αναμένονται και νέες θετικές εξελίξεις. Δηλαδή αυτές τις μέρες η Μακεδονία θα το, θα αλλάξει το γραφείο που διαθέτει στην Πρίστινα σε πλήρη πρεσβεία και ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και το κοσυφοπέδιο προς την Μακεδονία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο ερωτημάτων. Ο Στέφος ρώτησε για δύο λεπτά. Minister, it's good to see you in the, in the Foreign Affairs Committee Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ελπίζω το 2010 να είναι έτο επιτυχίας, όχι μόνο λόγω της άρσης της υποχρέωση θεώρησης, αλλά και λόγω της εκκίνηση των διαπραγματεύσεων, καθορισμού συγκεκριμένη ημερομηνία για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Τρία ερωτήματα, επιτρέψατε μου. Συμφωνώ ότι σχέση σας με την Ελλάδα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Θα μπορούσατε να μας πείτε πως εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να βρεθεί συμβιβασμός, διότι λύση σημαίνει συμβιβασμός ένθεν και ένθεν. Για την ονομασία του αεροδρομίου των Σκοπίων, δεν νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε μια χειρονομία καλής θελήσεως για να αλλάξετε το όνομα του αερολιμένος των Σκοπίων από πλευράς εσωτερικής κοινής γνώμης βεβαίως θα έχετε πρόβλημα. Το αναγνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ χρήσιμη χειρονομία καλής θέλησης να αλλάξετε το όνομα του αεροδρομίου των Σκοπίων. Με το Κόσοβο είστε θαραλέοι. Με τη Σερβία πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί, εις ό,τι αφορά την αναγνώριση και τα θέματα συνόρων, οι Σέρβοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη στάση σας. Τέλος. Βλέπω CNN και βλέπω διαφημίσεις. Επενδύστε στη Μακεδονία, λέει η διαφήμιση. Επενδύστε στη χώρα μας τι θα κάνετε για να προσελκύσετε ξένες επενδύσεις, ξένα κεφάλαια, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι είναι ζωτική σημασία για την ανάπτυξη της χώρας σας. Ευχαριστώ. Γκράτσιε. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ γκράτσιε. Ο κύριος Σαλαβράκος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Υπουργός, του οποίου διάβασα το βιογραφικό και είναι πάρα πολύ καλό, μίλησε με ηρεμία. Το βιογραφικό του μάλιστα εμπλουτίζεται και από το γεγονός ότι ε, υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κόκαλη, ενός μεγάλου ελληνικού ιδρύματος στο Χάρβαν, πράγμα που σημαίνει ότι οι Έλληνες στο πρόσωπό του έχουμε δείξει μια εκτίμηση και μια ιδιαίτερη κατανόηση. Όμως δεν θα μιλήσω σαν Έλληνα Ευρωβουλευτή. Θα θέλω να επισημάνω ότι οι λόγοι του κυρίου Υπουργού έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες θέσεις του Πρωθυπουργού της Φύρομ, ο οποίος επισκέφθηκε την Αυστραλία μέσα στο μήνα Οκτώβριο και μίλησε για Μακεδόνες του Αιγαίου που βρίσκονται στην Ελλάδα, Μακεδόνες του Πυρήν που βρίσκονται στη Βουλγαρία και Μακεδόνες της Βαρδαρίας που βρίσκονται στην Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας αντέδρασε άμεσα λέγοντας ότι η ΦΥΡΟΜ θέτει ζητήματα συνόρων με τη Βουλγαρία και ενώ παράλληλα η επίσης πρόσφατη οριοθέτηση των συνόρων ΦΥΡΟΜ Κωσόβου προκάλεσε αντίδραση του Βελιγραδίου. Είναι λοιπόν σαφές ότι σε διπλωματικό επίπεδο μέσα σε ένα διάστημα από 15 έως 31 Οκτωβρίου δύο γειτονικέ χώρες προς την ΦΥΡΟΜ εκτός της Ελλάδος, η Βουλγαρία και η Σερβία, ενοχλήθηκαν από τη συμπεριφορά της, αν δε σε αυτό συμπεριληφθεί και η εκκρεμότητα Ελλάδος Ελλάδος-Φύρων, αντιλαμβάνεστε ότι οι σχέσεις της χώρας αυτής, η οποία ευχόμεθα να, να βελτιωθεί σε σχέση με τους γειτονές της, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι τόσο καλή. Παράλληλα, σε οικονομικό επίπεδο, η χώρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση διότι ε, από ό,τι βλέπω έχει εγκριθεί για τη χρονική περίοδο 2009 έως 2013 ένα ποσό 494 εκατομμύριων ευρώ τα οποία δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που θα πάνε. Ερωτάτε λοιπόν, είναι διατεθειμένη η ΦΥΡΟΜ να επιδείξει μια μείωση της αδιαλαξίας της με τις γειτονικές χώρες και ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σαφω Πρέντα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την σημαντική πρόοδο που έχει επιτελέσει η ε, Μακεδονία για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ε, και για την καταπλέμιση της διαφθοράς. Στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, η εκκίνηση των ενταξιακών δραματευσεων αναφέρεται ως ένα πολύ σημαντικό κίνητρο που θα δώσει δυνατότητα στην πολιτική ελίτ να προβούν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ναι. ένταξη υπ' αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2009 θα πρέπει να επιβεβαιώσει αυτές τις συστάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να καθορίσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ε, θεωρώ ότι μια, ε, μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το σύνολο των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που έτσι θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτός ο οποίος πληρεί τα κριτήρια έχει μια ευρωπαϊκή προοπτική. Κύριε Υπουργέ, ένα ερώτημα προς εμάς. Αφορά το θέμα που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, το θέμα της διαφοράς με την Ελλάδα. Το ερώτημα που σας θέτω είναι το εξής. Ο καθορισμός μιας ημερομηνία για την εκκίνηση των διαπραγματεύσεων είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι διευκολύνει ή όχι την επίλυση της διαφοράς με την Ελλάδα. Θα ενθαρρύνει την εξέβρεση λύσης ή θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Μία ερμηνεία σας ζητώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα για δύο λεπτά η συνάδελφος Κορνέλισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πράσινοι πιστεύουμε ότι η κίνηση των πρώτων διαπραγματεύσεων για την Μακεδονία είναι θετικό. Είναι σημαντικό δε όχι μόνο για την Μακεδονία αλλά και για Άλλε υποψήφίε εν δυνάμει αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να επιβραβεύσουμε την Μακεδονία για την πρόοδο που επέτυχε και δεν θα πρέπει να μπλοκάρουμε το δρόμο της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λόγω διμερών διαφορών με άλλες ε, χώρες. Είναι ένα παράδειγμα που αφορά ε, την σχέση μας και με άλλες χώρες. Εσείς ε, κύριε Υπουργέ και η χώρα σας παρόλο ότι εργαστήκατε σκληρά και έχετε ήδη αποδώσει καρπούς δεν έχετε ακόμα επιβραβευθεί λόγω αυτής της διαφοράς. Από την άλλη, από την άλλη θα πρέπει βεβαίως να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της ονομασίας η ορμή που έχει αποκτηθεί σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διατηρηθεί. Πάντως εγώ θα ήθελα να θέσω ένα θέμα που αφορά τη διακριτική μεταχείριση και την καταπολέμηση αυτών των διακριτικών μεταχειρήσεων. Η έκθεση της Κομισιόν λέγει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος ε, για την οικιακή βία αλλά υπάρχουν ακόμα ανησυχίες για την πολιτική συμμετοχή των γυναικών, την εφαρμογή του νόμου για τις ίσες ευκαιρίες και ιδιαίτερα για τις διακριτικές μεχειρήσεις που υφίστανται οι σεξουαλικές μειονότητες που δεν την χάνουν καμία απολύτως προστασίας. Τι προτίθεστε να κάνετε στους τομείς αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κορνέλισεν. Ο κύριος ο Χουντής για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Υπουργό και τον ευχαριστώ πολύ. Για μας που προερχόμαστε από την Ελλάδα ήταν διπλά ενδιαφέροντα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται να υπάρχουν σχέσεις καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο λαών. Το παράδειγμα που αναφέρατε κύριε Υπουργέ ότι βρίσκονται στρατιώτε και από τι δύο χώρε για το Αφγανιστάν, εμένα με αφήνει αδιάφορο. Δεν έπρεπε να πάει κανένα, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Φύρο. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που μάλλον είναι στην ημερήσια διάταξη μετά. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα, και απευθύνομαι σε όλου του συναδέλφου, δεν είναι μια βαλκανική γραφικότητα το πρόβλημα του ονόματο, ούτε κάποια αιμονή ανεξήγητη. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, να λυθεί με τον καλύτερο τρόπο. Είναι αιστεία πιθανή ένταση στον χώρο των Βαλκανίων, δυσκολεύει να βοηθήσουμε όλοι μαζί αυτή η περιοχή να πάψει να αποτελεί αιστεία συγκρούσεων, εντάσσεων, να μπει σε έναν δρόμο ευημερία για το καλό των λαών και ούτω κάθεξης. Επομένω, πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατό, διότι τροφοδοτούνται εθνικισμοί εκατέρωθεν, θα πω. Δύο λοιπόν ερωτήσει. Από την πλευρά των περισσότερων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, εγώ προσθέτω τη φωνή του δικού μα χώρου, τη αριστερά, ενό κομματιού τη αριστερά, συμφωνούμε με αυτή τη σύνθετη ονομασία αμοιβαία αποδεκτή στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εδώ δεν δώσατε απάντηση, αν μπορείτε να πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο, κύριε Υπουργέ. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, είναι όλες οι δυνάμεις πολιτικές και πολιτιακές στη χώρα σας σύμφωνες με την τακτική της σημερινής κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα του ονόματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie, onorevole Ευχαριστώ κύριε Χούντι. Το λόγο έχει η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τον Υπουργό. Ε, θέλω όμως να σημειώσω ότι και σε αυτά που είπατε εσείς και άλλοι συνάδελφοι ε, ότι είναι περίπου μια αστεία υπόθεση το όνομα. Είναι σαν να λέτε στον Υπουργό ότι η χώρα του δεν πρέπει να κάνει απολύτω τίποτα για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα δεχτεί να μπει η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν δείξει ότι δέχεται αυτό ακριβώς που αποφασίστηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή να υπάρξει μια συνδιαλλαγή και μια συνεννόηση. Η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα αυτή προέρχονται από την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καλή είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά κάτω από τις γραμμές είναι ολοφάνερο ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα των ατομικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των διαφόρων ομάδων, ότι η θέση των γυναικών είναι τραγική, ότι η διαφθορά είναι μεγάλη, ότι υπάρχει τράφικινγκ γυναικών. Και ακόμη, κάτι που δεν φαίνεται σαφώς στην έκθεση της Επιτροπής, ότι υπάρχουν εθνικιστικές κραυγές από την πλευρά της κυβέρνησής σας, κύριε Υπουργέ. Τα σχολικά σας βιβλία περιλαμβάνουν απίστευτη προπαγάνδα με αναφορές στους γείτονες. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι η χώρα σας απειλεί την Ελλάδα, δεν μπορεί να την απειλήσει. Εκ των πραγμάτων δεν είστε σε θέση να απειλήσετε την Ελλάδα και επομένω δεν την απειλείτε. Εγώ λέω ότι παραδείγματο χάρη μεγαλώνεται μια νέα γενιά πολιτών με εμπάθεια, εθνικισμό και φοβερή προπαγάνδα. Τα σχολικά σας βιβλία τα γνωρίζω καλά γιατί υπήρξα υπουργό Παιδείας και θέλω να μου απαντήσετε από αυτού. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Γιαννάκου. Το λόγο έχει ο κύριος Κύριλοφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η απάντηση είναι, η απόφαση είναι καλή όσον αφορά την κατάργηση των θεωρήσεων. Αλλά σωστά τα, οι νέοι διαβάζουν αυτά τα σχολικά βιβλία που δημιουργούν μίσος εναντίον των γειτόνων. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν ότι οι γείτονε είναι καλοπροαίρετοι. Επίση, όσον αφορά τις ε, εξελίξεις, ε, όντως ε, έχετε πάει καλά κύριε Υπουργέ, αλλά έχω να κάνω μία ανθρώπινη ερώτηση. Με τους συναδέλφους του ΕΛΚ αποφασίσαμε πριν λίγο καιρό να ε, επισκεφθούμε ε, βουλγαρικά μνημεία στα σύνορα και τρομάξαμε δεν μπορούσαμε όμως να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας στον τύπο σας. Συναντήσαμε ε, του υπουργούς. Είναι μια πολύ ανθρώπινη ε, υπόθεση διότι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να επισκεφθούν τα μνήματα των οικογενειών τους. Υπάρχουν ιδίως ε, δύο-τρεις περισσότερες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να επιληθούν σε δύο-τρεις εβδομάδες. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να λήξετε ε, όλα τα θέματα. Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Μποτσεύσκη μετά παρετήθηκε από αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά εσείς είσαστε εδώ. Λοιπόν, γιατί δεν ε, επιτύχατε. Μας είχατε πίσω όταν σας συναντήσαμε, ήταν πολύ φιλική η συνάντηση. Κάτι μας υποσχεθήκατε, το οποίο όμως δεν σεβαστήκατε. Για εξηγήστε μας παρακαλώ τι συμβαίνει. Ευχαριστώ κύριε Κύριλοφ. Το λόγο έχει η κυρία Βάγγελ για δύο λεπτά. Ο κύριος Βάγγελ. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που είστε εδώ και χαίρομαι που το μέλλον σας είναι συνδυασμένο με ε, σαφείς επιτυχίες στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Ελπίζω να είναι συνδεδεμένο επίσης με ε, παραδοσιακές ε, φιλικές σχέσεις τις οποίες εσείς πρεσβεύετε. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ ιδίω ε, εφόσον έχουμε ανοίξει την πόρτα για τη νεολαία για να διακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημερινή συζήτηση πήγε, πάει προς σωστή κατεύθυνση διότι αποδεικνύει ότι έχει διαφανεί σαφώς ότι ε, για τη Μακεδονία, για τη Φύρομ είναι πιο βασικό το μέλλον από ότι το παρελθόν. Το παρελθόν είναι πάντοτε σημαντικό, αλλά το παρελθόν δεν πρέπει να αποτελέσει το στοιχείο το οποίο εμποδίζει ένα κράτος να ε, μετεξελιχθεί σε μία σύγχρονη κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να απαρνηθείτε τον ιστορικισμό να γίνεται ένα πραγματικά σύγχρονο κράτος το οποίο ε, θα βρει μια κοινή δυνατότητα ε, συζητήσεως με τους γειτόνους σας. Αυτή είναι προτεραιότητα, ιδίως για νέους ανθρώπους όπως και εσείς και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για την ε, αλληλεγγύη την οποία έχετε επιδείξει και ιδίως για την ε, θέση σας κατά την κρίση του Κωσυφοπεδίου. Ο κύριος Πέτερλε τώρα. Ευχαριστώ ή πάντοτε πίστευα ότι είναι πολύ σημαντικό να προσχωρήσει η ε, ΦΥΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χαίρομαι για τις πρόοδους που έχετε κάνει και ε, θα χαιρετίζω και την αισιοδοξία σας για το μέλλον. Ελπίζω ότι δεν θα, υπάρξουν, ε, ε, δεν θα υπάρχουν προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση και το εύχομαι και για μας και για την ε, χώρα σας. Χαίρομαι για αυτό που μας είπατε για την οικονομία και την κατάστασή της στη Μακεδονία ε, χαίρομαι ε, για το, το θάρρος ε, το οποίο επιδείξατε και χαίρομαι για την ελεύθερη διακίνηση ατόμων ξέρω ότι εύχομαι ότι σύντομα θα μπορούμε να ε, καλωσορίσουμε πολλούς από τους συμπολίτε σας στην Ευρώπη. Ε, ελπίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα με την Ελλάδα, ότι θα κάνετε κινήσεις που θα επιτρέψουν να επιληθούν τα ακόμη ανοιχτά προβλήματα. Γι' αυτό και θα έλεγα να υπάρξουν και άλλες κινήσεις σαν αυτό το άνοιγμα του σταθμού των ε, συνόρων. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε επίσης συνεργασία με τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Μακοβέη για δύο λεπτά. Η κυρία. Θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι έχω εργαστεί δύο χρόνια στα Σκόπια, 2007-2008 και ε, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουν υπάρξει πρόοδοι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σας κυρία μου. Μπορείτε παρακαλώ να πλησιάσετε στο ένα μικρόφωνο το οποίο λειτουργεί. Ευχαριστώ. Τώρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι δύο χρόνια ε, εργάστηκα το 2007-2008 ε, στη ΦΥΡΟΜ σαν μέλος της ε, της ε, πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου να στηρίξουν ε, την περιοχή ε, και είδα την καταπολέμηση της διαφθοράς, της κατασχέσεις στο νέο ποινικό δικαστήριο το οποίο έχει καταρτιστεί, την νομοθεσία η οποία έχει υιοθετηθεί και ε, πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνονται ίσως όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή ότι όλες οι δικαστικές αποφάσεις δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα, ε, ότι έχει οθετηθεί ε, μία προσπάθεια διαφάνειας. Είδα λοιπόν και τις προσπάθειες και τις δυνατότητες του λαού αυτού να αποδώσει και θέλω να ενθαρρύνω αυτή τη χώρα στις προσπάθειες να τη συγχαρώ και να της πω ότι ελπίζω ότι θα επιβεβαιωθεί η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι σημασία έχουν τα επιτεύγματα της χώρας σε αυτό το θέμα. Εάν λοιπόν δούμε ποια είναι τα προσόντα και τα επιτεύγματα, ελπίζω ότι θα υπάρξει μία απελευθέρωση των ε, ε, θεωρήσεων και ότι θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, τον Ιανουάριο του 2010. Ε, πρέπει επίσης να λυθεί το θέμα της ονομασίας χωρίς να θέλουμε να τιμωρήσουμε το λαό ο οποίος εργάστηκε σκληρά. Δεν θα ήταν σωστό και γι' αυτό εμείς είμαστε υπέρ της ισότητος και τέλος Πιστεύω ότι ε, ε, για, σαν αναγνώριση των προσόντων ε, θα μπορέσουν να προχωρήσουν με τις διαπραγματεύσεις και τα θέματα της ονομασίας διαφορετικά θα υπάρχει αδικία η οποία δεν θα βοηθήσει την, τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ την κυρία Μακοβέη. Τα, τα, ε, τις παρεμβάσεις θα ολοκληρώσει ο κύριος Κουμουτσάκος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μαζί με άλλους ε, συναδέλφους και εγώ βλέπω ότι η χώρα σας έχει κάνει μια θετική στρατηγική επιλογή να γίνει μέλος ευρωπαϊκής οικογένειας και ό,τι πρόοδο έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ την καλωσορίζω. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι ενώ στο εσωτερικό γίνονται πραγματικά ειλικρινείς προσπάθειες μεταρρυθμίσεων προς σωστή κατεύθυνση, στο πεδίο των σχέσεων καλής γειτονίας έχουμε μια ανάστροφη πορεία. Επί ημερών της κυβερνήσεως που συμμετέχετε, της κυβερνήσεως Γκουρεύσκη, έχει σαφώς σημειωθεί μια τάση χειροτέρευσης των σχέσεων της πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας και με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία, δύο, γειτονικά σας κράτη που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση είναι τι θα κάνετε για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Και θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλές ενέργειες που έχουν γίνει και θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει για να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ της χώρας σας και των γειτονικών της χωρών. Θα επιμείνω μόνο σε ένα. Θα ανασταλεί η έκδοση χαρτών που δείχνουν την ύπαρξη μιας μεγάλης Μακεδονίας με εδάφη της Ελλάδας μέχρι και τη Θεσσαλονίκη αλλά και της Βουλγαρίας. Ε, κύριε Υπουργέ, η ατμόσφαιρα ανυφαλιότητας και ηρεμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε διαπραγμάτευση. Και βεβαίως αυτό απαιτείται και για την τρέχουσα διαπραγμάτευση στον, ε, στα Ηνωμένα Έθνη. Είστε έτοιμοι να αποδεχτείτε το συμβασμό που προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για ένα όνομα, το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ώστε να μην υπάρχει μονοπόληση του ονόματος μιας ολόκληρης περιοχής. Για φανταστείτε τη Σκανδιναβία, αν στη Σκανδιναβία που αποτελείται από τη Δανία, τη Σουηδία, την Νορβηγία, ένα από αυτά τα τρία κράτη να ονομαζόταν ξαφνικά Σκανδιναβία και να νόμιζε το λαό της Σκανδιναβούς και τη γλώσσα Σκανδιναβική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκη. Έχετε πολλές ερωτήσεις κύριε Υπουργέ και λίγο χρόνο και ε, σας εύχομαι καλή τύχη για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα σχόλια, λέγει ο Υπουργός. Ε, ε θέλω να πω στους ε, ε εκπροσώπους εδώ ότι ε, χαιρόμαστε που μπορούμε να ε, ε, ε, συζητήσουμε στην ουσία το θέμα της περιοχής. Και κύριε Κουμουτσάκη, θέλω να σας πω ότι η χώρα μας είναι ένα νέο σύγχρονο κράτος ειρηνικό που ενδιαφέρεται να αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους γειτονές της και που ενδιαφέρεται για την ευημερία της χώρας μας, των γειτόνων και της περιοχής. Θα ήθελα να ε, υπενθυμίσω στο κοινό ότι τον Ιανουάριο Ιανουάριο 2008, δηλαδή λίγο πριν από τη διάσκεψη κορυφής του Βουκουρεστίου, η ΦΥΡΟΜ είχε παραστεί σε μία συζήτηση ε, στη Διοχρίδα με τον πρέσβη Βασιλάκη και τον πρέσβη Δημήτροφ εκείνη την περίοδο και είχα δώσει ένα σχέδιο κοινού ψηφίσματος το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει τους Έλληνες συναδέλφους μας και μιλούσα για συνεργασία, για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της, ε, της εταιρικής σχέσεως. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με αμοιβαίο σεβασμό. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει και όχι να μπλοκάρει τη την προσχώρηση της περιφέρειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε μία αθρώα προσέλευση Ελλήνων επιχειρηματιών στη χώρα μας, άρα έχουμε περισσότερα κοινά σημεία παρά διαφορές. Επίσης, ε, ε, η Ελλάδα είναι η χώρα που επισκέπτονται οι περισσότεροι υπήκοοι της χώρας μου, άρα σε επίπεδο επίπεδο κατοίκων υπάρχουν πιο πολλοί δεσμοί και κύριε Μουτσάκο, εσείς και εγώ ίσως ε, έχουμε συμβάλει ε, σε αυτήν την δυσάρεση κατάσταση αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να, να αξιολογήσει κάποιος άλλος τα θέματα αυτά πιο αντικειμενικά. Στην κυρία Μακαβέη την ευχαριστώ ε, για την ε, συνδρομή της ε, για τα συγχαρητήριά της για τον αγώνα μας κατά της κατά της διαφθοράς και είμαστε πολύ ευτυχής για την πρόοδο ε, η οποία αναγνωρίζεται ε, για τα επιτεύγματα της χώρας μας. Ελπίζουμε ε, ότι είμαστε ειρηνικοί και ότι θα το αποδείξουμε και στο μέλλον. Όσον αφορά τον κύριο Πέτερλε, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Όσον αφορά την αρχική μας ε, πρωτοβουλία που θα μπορούσε ε, ε, να είναι προς όφελος της περιοχής και της χώρας μου, θέλω να τονίσω ότι εμείς την χάνουμε